Πριν ξεκινήσουμε τις εργασίες ε, της σημερινής Ολομέλειας, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τα θύματα των πυρκαγιών στα δάση που, έγιναν, που έλαβαν χώρα στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, τις τελευταίες εβδομάδες. Όπως είχα πει και στην παρέμβασή μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το φαινόμενο είναι ανησυχητικό και αξίζει της προσοχής μας. Μόνο φέτος στην Ευρώπη 750.000 εκτάρια δασών καταστράφηκαν φέτος και μόνο στην Πορτογαλία 100 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Γι' αυτό λοιπόν είμαι πεπισμένος ότι είναι και η ώρα να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό σώμα προστασίας και να πλουστεύσουμε το νομοθετικό πλαίσιο, τόσο ώστε να επιτρέψουμε στου πληθυσμού να λάβουν άμεση βοήθεια σε περίπτωση που τη χρειάζονται. Σας ενημερώνω επίσης για την απόφαση που λάβαμε με κοινή συμφωνία με τον πρόεδρο Τούσκ και τον πρόεδρο Γιούνκερ να δώσουμε στους πληγέντες από τις πυρκαγιές των δασών το ποσό που λάβαμε από το, τους πρίγκιπες της Αστούριας στα πλαίσια του βραβείου που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση την περασμένη Παρασκευή στο Βιέδο. Το ποσό αυτό που λάβαμε θα το δώσουμε στους ε, πληγέντες. Με αυτόν τον τρόπο θα δείξουμε την αλληλεγγύη μας ε, προς, τους, προς τα θύματα και προς τα, τις οικογένειες των θυμάτων στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Για αυτά τα θύματα θα ήθελα να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή κατά τη διάρκεια του οποίου θα τιμήσουμε και τα θύματα της Ιρλανδίας ε, του τυφώνα Οφιλία. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αύριο, πριν την ψηφοφορία, θα τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή για να τιμήσουμε τη Μαλτέζα δημοσιογράφο Ντάφνε Γκαλουάνα Γκαλίσια που δολοφονήθηκε σε μια απόπειρα κατά τη ζωή της την περασμένη εβδομάδα. Θα κάνουμε μια πολύ σύντομη τελετή αύριο Αύριο θα είναι παρόντα στην Ολομέλεια και τα μέλη της οικογένειάς της. Τα προσκαλέσαμε, δέχτηκαν την πρόσκληση και θα παραστούν ε, στην, στις θέσεις εδώ της Ολομέλειας. Στα θεωρία της Ολομέλειας.